Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώς ήρθατε στην απογευματινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης. Δεν ήταν δύσκολο να βρείτε την αίθουσα, στη διπλανή μεταφερθήκαμε. Είχα την εντύπωση κιόλας ότι το πρωί είχαμε περισσότερη λιακάδα. Λοιπόν, συνάδελφοι, πριν το μεσημεριανό διάλειμμα ανακοινώσαμε μια αλλαγή στην ημερήσια διάταξη και ευχαριστώ πάρα πολύ τη Λόλα η οποία μας επέτρεψε να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη. Σημείο 23 θα το εξετάσουμε τώρα αντί για το σημείο 21, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε για την τρίτη διεθνή διάσκεψη για την ανάπτυξη. Είχαμε στείλει μια αντιπροσωπεία εκεί. Η συνεδρία ήταν ιδιαίτερα σημαντική, διότι το θέμα ήταν πώ θα βρούμε τα κονδύλια για να χρηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη, κάτι που θα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Πέντρο Σίλβα Περέιρα είναι ο εισηγητή, ήταν μαζί μα και θα μα παρουσιάσει την ε, το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να συμμεριστώ τα αποτελέσματα της ε, συνδιάσκεψης στην Αντίσα Μπέμπα για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Η πρώτη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι η εξής. Υπήρξε συμφωνία στην Αντίσα Μπέμπα, εγκρίθηκε ένα έγγραφο, μια ημερήσια διάταξη, ένα θεματολόγιο δράσης που είναι γνωστό ως θεματολόγιο δράσης της Αντίσα Μπέμπα και θα είναι ένα μέσο υποστήριξης στην εφαρμογή της ε, ημερήσιας διάταξης για την ανάπτυξη μετά το 2015 που θα συζητήσουμε τώρα και στην επόμενη συνδιάσκεψη της Νέας Υόρκης. Αυτό το έγγραφο δεν είναι λοιπόν όλα, δεν είναι το σύνολο εκείνων που επιθυμούμε. Και νομίζω ότι μπορώ να πω ότι δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο είναι το αναγκαίο ιδιαίτερα για τα πιο σημαντικά θέματα και είναι για τις δεσμεύσεις τις χρηματοοικονομικές, τις συγκεκριμένες και χειροπιαστές που απαιτούν προσθήκες και πρόσθετα κονδύλια για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της ανάπτυξης. Είναι ένα θεματολόγιο για την ανάπτυξη χωρίς εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη. Αυτό είναι όλο και όλο. Και αντιβαίνει στη φιλοδοξία αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλων εκείνων που επιθυμούσαν να έχουμε μια διάσκεψη μεγάλων φιλοδοξιών και προσδοκιών για να λειτουργήσουν οι στόχοι για την ανάπτυξη που επιθυμούσαμε. Πρέπει να αναγνωρίσω όμως ωστόσο ότι πολλές από τις συστάσεις μας και διεκδικήσεις μας συμπεριλαμβάνονται στο τελικό έγγραφο που είναι ένα έγγραφο πολύ ολοκληρωμένο θα έλεγα και καλύπτει όλους τους μεγάλους τομείς από τις, ε, τους πόρους ε, και για το θέμα της διεθνούς χρηματοδότησης επίσης την διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη, το εμπόριο, μία αναφορά με με τριόφρονα για το θέμα της αηφορίας, της βιωσιμότητας των, του δημοσίου χρέους και μετά θέματα που αφορούν την επιστήμη, την τεχνολογία, την ανάπτυξη, την κατάρτιση και εκπαίδευση επαγγελματική και την ενίσχυση του δυναμικού των κρατών μελών για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις για την ανάπτυξη. Για όλους αυτούς τους λόγους, σε ένα τόσο μεγάλο ευρύ έγγραφο, με τόσο ευρύς ορίζοντες είναι εύκολο να βρει κανείς διάφορα κεφάλαια στα οποία μπορεί κανείς ε, να αποτυπώσει ή να δώσει τις διαστάσεις ε, των οραμάτων μας, του ονείρου μας για την καταπολέμηση της φτώχειας και την επίτευξη μιας αηφόρου ανάπτυξης. Ωστόσο, όπως είπα, αυτό το έγγραφο δεν πετυχαίνει αυτό που είναι αναγκαίο για συγκεκριμένες αποφάσεις. Δεν υπάρχουν νέες δημοσιονομικές δεσμεύσεις για κονδύλια επιπρόσθετα. Και για την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο εκείνη τόνισε τους στόχους αυτούς και που πρέπει να επιτευχθούν. Κανένας άλλος από τους διεθνούς εταίρου, διεθνείς εταίρους δεν το έκαναν. Και υπάρχει μια παράγραφο στο τελικό έγγραφο που ακριβώς δίνει τη διάσταση αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι ξεχώρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο μόνο διεθνής εταίρο που δεσμεύτηκε με τους στόχους αυτούς και για το τέλος της περίοδου μέχρι το 2030 να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Άλλα θέματα θα μπορούσαν να είναι μια μεγαλύτερη ανάπτυξη. Η συζήτηση όμως επικεντρώθηκε στο θέμα, στο θέμα του οργάνου, του μέσου των Ηνωμένων Εθνών για την ε, δημοσιονομική συνεργασία ε, επικεντρώθηκε η συζήτηση τι θα μπορούσε να γίνει διακυβερνητικά με ένα όργανο ή αν θα είχαμε ένα τεχνικό όργανο μεταξύ των κρατών μελών κάτι το οποίο σε σχέση με τις απαιτήσει ε, δεν είναι ίσως το πιο ενδεδειγμένο. Εδώ βλέπουμε και μια μεικτή ε, προσέγγιση. Δεν έχουμε ούτε διακυβερνητικό όργανο, αλλά υπάρχει μια πιο δραστήρια συμμετοχή των κυβερνήσεων στην επιλογή των ε, στοιχείων που θα συναποτελούν αυτό το όργανο συνεργασίας. Και πάλι εδώ δεν είχαμε μια λύση μεγάλων τροποποιήσεων σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο υπήρξε σαφώς ε, απουσία φιλοδοξιών όσον αφορά τη νέα εμπλαισίωση, το νέο πλαίσιο σε ε, διεθνή κλίμακα για τα ε, δημόσια χρέη. Και η περίπτωση της Αργεντινής δείχνει ότι κάτι τέτοιο είναι απόλυτο αναγκαίο να γίνει. Και μετά για τον ιδιωτικό τομέα που όλοι μας θα θέλαμε να βλέπαμε καλύτερες εγγυήσεις και εχέγγυα για την ευθυγράμμιση και τη συμμόρφωση του ιδιωτικού τομέα για την ε, αϊφόρο βιώσιμη ανάπτυξη. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με μια παρατήρηση που έχει πολιτικό χαρακτήρα όσον αφορά τη διεθνή κοινότητα και την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Είναι παράξενο, είναι αξιοπερίεργο <clears throat> ότι το 0,7% η δημόσια χρηματοδότηση για την ανάπτυξη δεν βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των συζητήσεων και ο κύριος λόγος πιστεύω εγώ γι' αυτό και σε σχέση με την αντιπροσωπεία μας που παρακολούθησε αυτές τις αντιπροσωπίες, ε, αυτές τις διαπραγματεύσεις είναι ότι ακόμα και στην ομάδα που ενδιαφέρεται περισσότερο για αυτό το θέμα της, ε, του, της ομάδας ε, των 7 των αναδειωμένων κρατών επικαλύπτεται η προσπάθεια αυτή και επικαλύπτει τις προσπάθειες των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και έτσι λοιπόν δεν ενδιαφέρει πλέον κανέναν αυτό το θέμα. Ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μπόρεσε να πάει πιο πέρα με μια θέση μεγάλων φιλοδοξιών. Σίγουρα όχι με τις ε, ε, χώρες που δεν θέλουν να υπομισθούν περισσότερες δεσμεύσεις. Ούτε για τις αναδυόμενες ε, οικονομίες που μια σημεριζόμενη ευθύνη θα σήμαινε αυξημένες ευθύνες και για αυτές τις αναδυόμενες οικονομίες. Και οι μόνοι ενδιαφερόμενοι ποιοι είναι οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες που έχασαν τη φωνή, δηλαδή δεν μπόρεσαν να επιβάλλουν τις θέσεις τους και σε σχέση με την ευρύτερη ομάδα. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται αυτή η διάσκεψη και στο τέλος του εγγράφου βλέπουμε αυτά τα στοιχεία. Όμως δεν μπορούμε να κρίνουμε ότι δίνονται εχέγγυα μεγάλης επιτυχίας για την επίτευξη της αηφόρου της βιώσιμης ανάπτυξης που θέλουμε να προωθήσουμε. Έτσι προχωρούμε λοιπόν για τη διάσκεψη της Νέας Υόρκης και τη διάσκεψη των Παρισίων. Διαρκώς αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα, που είναι το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και με το θέμα των προσφύγων. Πάρα πολλές συζητήσεις, πολιτικά θέματα, ε, ε, έγγραφα που εγκρίνονται, ωστόσο δεν υπάρχουν δεσμεύσεις για να μπορέσουν να αλλάξουν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις για τον Πέδρο.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 Ναι, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δυστυχώς δεν είναι εδώ για να απαντήσει την ερώτησή σας, όμως σίγουρα είναι μια ερώτηση που πρέπει να γίνει, διότι διαφορετικά δεν θα δούμε χρηματοδότηση. Propose un débat au Parlement public, au Parlement européen en séance plénière. Il faut plus se cacher derrière son petit doigt, il faut que les engagements pris soient tenus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 να βάλουμε ως ύψιστη προτεραιότητα την παρακολούθηση της εγκατάσταση μετά την Αντισαμπέμπα, διότι πρέπει να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει και αυτή ευθύνη. Από όσο ξέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει μια ξεχωριστή έκθεση σχετικά με την κινητοποίηση των εγχώριων ε, πόρων για την ανάπτυξη. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα στοιχεία που συνθέτουν την όλη εικόνα. Εμείς πρέπει να ασκήσουμε πίεση έτσι ώστε να διασφαλίσουμε το ότι θα γίνουν ενέργειες. Και αυτό θα συζητηθεί αργότερα με τους ε, συντονιστές. Θα υπάρχει λοιπόν παρακολούθηση και θα το συζητήσουμε. Όντω χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα εργασία, διότι αν περιμένει ε, για πέντε χρόνια δεν θα γίνει τίποτα. Η αναμονή δεν οδηγεί σε αποτελέσματα. Χρειάζεται πίεση έτσι ώστε να κινηθούν τα πράγματα. Και αυτό ήταν ένα από τα ενδιαφέροντα θέματα στην Αντισαμπέμπα ε, για τις ε, χώρες που έχουν περισσότερη ανάγκη, η αναπτυξιακή βοήθεια είναι ύψη της σημασίας. Για τις αναπτυσσόμενες είναι λιγότερο. Η περίπτωση της Νιγηρίας για παράδειγμα, σε σύγκριση με την ε, περίπτωση του Μάλι, μα ε, δείχνει αυτό το θέμα. Το Μάλι είναι από τι ε, πιο φτωχέ χώρε τη Αφρική και η αναπτυξιακή βοήθεια έχει όντω μεγάλη σημασία και παίζει ρόλο. Εάν δεν υπάρχουν λοιπόν άλλα σχόλια, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πέδρο, να ευχαριστήσω και την Λόλα για την ευελιξία που έδειξε και νομίζω πως τώρα έχουμε χρόνο να περάσουμε στο σημείο 21 το οποίο αφορά την εφαρμογή των συστάσεων του Κοινοβουλίου του 2010 σχετικά με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική ευθύνη. Είναι μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με μια γνωμοδότηση που συντάξαμε για την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Ε, είναι παρόμοιο με το θέμα που είχε αναλάβει ο Σάρλ την ε, προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία και τώρα θα δούμε αν υπήρχε συνεκτική πολιτική για την ανάπτυξη και μπορείτε να μας παρουσιάσετε τη γνωμοδότηση τώρα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Λίντα. Εμείς πιστεύουμε ότι η ευθύνη και η λογοδότηση σε σχέση με τις ε, ιδιωτικές επιχειρήσεις για τις δράσεις τους είναι θεμελιώδες στοιχείο και είναι ένα στοιχείο διαφάνειας και δημοκρατικότητας, δηλαδή κανείς να μην μπορεί να παραβαίνει τον νόμο. Για μας είναι απαράδεκτο πώς υπάρχει ατιμορρησία σε σχέση με αυτά τα θέματα και ζητούμε να υπάρχουν εγγυήσει για τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα για τα, τις γυναίκες, τα κορίτσια, τα παιδιά που εργάζονται πολλές φορές υπό όρους δουλείας, σκλαβιάς καθώς επίσης και για το περιβάλλον που είναι δημόσιο αγαθό και είναι αναγκαίο αγαθό για την επιβίωσή μας. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν η αναγκαία προστασία. Πρέπει να προστατέψουμε τους ανθρώπους για οποιαδήποτε παραβίαση των πιο θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Το πρώτο που πρέπει να απαιτηθεί είναι σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμάς τους ίδιους είναι να είμαστε συνεκτικοί και ε, να υπάρχει συνεκτικότητα και συνάφεια με τις πολιτικές μας όσον αφορά και τις συνθήκες Λισαβόνας και τη δράση μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δίνει με το ένα χέρι για την ε, διεθνή συνεργασία και την ανάπτυξη και να παίρνει με το άλλο χέρι με τις εμπορικές συμφωνίες που υπογράφουμε με αυτές τις χώρες. Πρέπει να διασφαλιστεί το ε, δικαίωμα για την ανάπτυξη που είναι αναφέρετο δικαίωμα, αναπαλωτρίωτο δικαίωμα όλων και γι' αυτό είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να σέβεται τα κυρίαρχα δικαιώματα των εθνών και των λαών και να θεσπίζονται πολιτικές που ανταποκρίνονται στα συμφέροντα των πολιτών και όχι τα συμφέροντα των επιχειρήσεων. Και όταν θέλουμε να έχουμε τα περιβαλλοντικά θέματα πρέπει να υπάρχει κοινή ευθύνη αλλά διαφοροποιημένη ευθύνη. Δεν έχουμε όλα τα κράτη τις ίδιες ικανότητες και δυνατότητες να αντιμετωπίσουμε περιβαλλοντικά θέματα και ούτε έχουμε και τις ίδιες ευθύνες. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι έχουμε ιστορική ιστορικέ ευθύνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το υπόλοιπο τη οικουμένη των άλλων κρατών του πλανήτη. Πρέπει να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια για τι δράσει των επιχειρήσεων. Δεν μπορεί να υπάρξει λογοδότηση για τα πεπραγμένα χωρί διαφάνεια και πρέπει να υπάρχει μελέτη επιπτώσεων εξ άντε, εκ προηγουμένου δηλαδή, εκ προημίου και να δούμε τι θα γίνεται σε σχέση με τις επιχειρήσεις που εποφελούνται από τις εμπορικές συμφωνίες που υπογράφουμε με τρίτες χώρες. Πρέπει να έχουμε ένα δεσμευτικό πλαίσιο ρυθμιστικό, δεσμευτικό για την, τον σεβασμό των κοινωνικών δικαιωμάτων, περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και ανθρώπινων δικαιωμάτων, διότι οι ρήτρες που υπάρχουν στις εμπορικές συμφωνίες μας σήμερα για αυτά τα δικαιώματα δεν είναι δεσμευτικές και πρέπει διαρκώς να επαγρυπνούμε για την υλοποίηση και εφαρμογή αυτής της ρήτρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη πιστεύουμε ότι πρέπει ενεργά να εμπλακούν σε σχέση με τα Ηνωμένα Έθνη και μέσω μιας διεθνούς συνθήκης, ώστε να υπάρχει ευθύνη και λογοδότηση για τις πολυεθνικές εταιρείε σε περίπτωση παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και περιβαλλοντικών διατάξεων. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στη γνωμοδότησή μας και ελπίζω ότι όλοι θα υπερψηφίσουμε και θα κινηθούμε προς την ίδια κοινή κατεύθυνση, διότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανάπτυξης πρέπει να είναι ενωμένη σε αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Σάντσες Καλέντε. Ο κύριος Κόζα έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚ. κυρία Κόζα. Habitához,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 γιατί μιλάμε για την πολιτική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται την κυριαρχία των ε, υποανάπτυξη χωρών. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς όπου θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα που θα μπορούσε να ε, έχει μεγαλύτερη συμμετοχή, αποτελεσματικότερη συμμετοχή στους στόχους ανάπτυξης. Ό,τι αφορά τους στόχους ανάπτυξης θα πρέπει να πούμε ότι είναι σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό και σε επίπεδο περιβαλλοντικό λαμβάνουμε υπόψη μας τα όσα μας περιβάλλουν. Πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Γι' αυτά είναι υπεύθυνα υπεύθυνε σε ενδιαφερόμενες χώρες, οι εμπλεκόμενες χώρες. Θα πρέπει να δούμε οι εμπλεκόμενες χώρες να παρέμβουν με τρόπο ενεργό στην ανάπτυξή τους. Θα επιθυμούσα οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες που πρόσφατα συμπεριέλαβαν ε, ρήτρες που αφορούν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ελπίζω λοιπόν τα έγγραφα αυτά να μας επιτρέψουν να επιτύχουμε μια πιο αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων. Εγώ θα υποβάλω τροπολογίες που επιτρέπουν να δοθεί μια πιο θετική χρειά και θα επιτρέψουν να υιοθετήσουμε μια πιο θετική προσέγγιση του θέματος. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε στην περιοχή ίντε προτάσεις που θα μπορούσαν να δείξουν τους στόχους της ανάπτυξης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων και είμαι στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία. Thank um, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ καλωσορίζω τη γνωμοδότηση από τη συνάδελφο Σάντσες. Πιστεύω πως είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή, μια πολύ καλή αφετηρία για την εφαρμογή των συστάσεων του 2010 για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ε, εταιρική ευθύνη. Κυρίε και κύριοι, οι εμπορικές μας πολιτικές πρέπει να αποτελέσουν εργαλείο για την προώθηση όχι μόνο των εμπορικών συμφερόντων μας, αλλά επίσης και να γίνει ένα μέσο που θα εφαρμόσει στην πράξη τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε στενότερα την εφαρμογή τους, έτσι όπως προβλέπεται από τις συνθήκες. Επίσης, ε, στηρίζω την ε, στήριξη των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη και να δημιουργηθεί η δυνατότητα να υπάρχει λογοδοσία από τις επιχειρήσεις για, το, ε, για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ενεργειών τους. Τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά και πρέπει να είναι μια υψηλότερη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα ε, για την εξάλληψη της φτώχειας. Εάν οι πολιτικές μας δεν είναι συνεκτικέ, τότε δεν θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε την ανάπτυξη και θα καταλήξουμε να δαπανίσουμε περισσότερα κονδύλια από ό,τι χρειάζεται. Η αναπτυξιακή βοήθεια έχει πλέον στις μέρες μας γίνει θέμα των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ορισμένα ζητήματα όμως είναι υπερβολικά σημαντικά για να τα αφήσουμε στα χέρια της αγοράς. Πρέπει οι καταναλωτές να ζητήσουν την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Συνεπώς η ευθύνη των πολιτών για τη συμφωνία αυτή είναι να διασφαλίσουν ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν θα έχει ως ε, συμφέρον μόνο τα οικονομικά ε, ωφέλη αλλά και τα ωφέλη των πολιτών. Αυξάνοντας τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα θα διασφαλίσουμε την ε, αηφορία των χωρών και την παραγωγικότητά τους. Χρειάζονται περιφερειακές και διμερείς συμφωνίες. Δυστυχώς, αυτήν την στιγμή έχουμε παρακολουθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποδειχθεί αδύναμη στις διαπραγματεύσεις. Πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειάζεται να ενισχύσουμε τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες έτσι ώστε να μπορέσουν να οικοδομήσουν την οικονομία τους. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να ε, ασκηθεί πίεση έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι διατάξεις της ε, συμφωνίας. Τέλος κυρίε και κύριοι, η κοινωνική εταιρική ευθύνη είναι κάτι που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε. Πολλές επιχειρήσεις ε, μας στήριξαν για τη δημιουργία υποχρεωτικής νομοθεσίας, όμως καταφέραμε παρόλες τις αντίξωες συνθήκες να ψηφίσουμε για τα περαιτέρω βήματα και πιστεύω πως μόνο μία συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα οδηγήσει αποτελέσματα. Και ελπίζω ε, όλοι οι συνάδελφοι να στηρίξουν τις τροπολογίες που θα υποβάλω. Ευχαριστώ πολύ. Σουάλ δεν σας είδα, θα σας δώσω το λόγο. Σας παρακαλώ, συνάδελφοι, να είστε σύντομοι, διότι μετά θα έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σουάλ, Μαρία και μετά η Χέντι. Δύο πράσινε στη σειρά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ την κυρία Σάντσες για αυτό που έκανε. Το ερώτημα είναι πώς, τι θα πρέπει να κάνουμε με βάση τις υποδείξεις της. Καταρχάς διαπιστώνουμε ότι στην Ευρώπη είναι αδύνατο να υπάρξουν νόματα σε όλες ε, τους ε, τομείς. Υπάρχουν ε, διατάξεις που διέπουν τις κοινωνικές πτυχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένες χώρες έχουν opt-out. Το θέμα είναι, δεν είμαστε πλέον σε θέση να επιβάλλουμε προς τα έξω αυτό που θέλουμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα που θέτω συνεπώς είναι με τι τρόπο θα επιβάλλουμε τι είδους πρότυπα. Στην περίπτωση, στα πλαίσια των διεθνών εμπορικών συμφωνιών παραμένει μία δυνατότητα να συμπεριλάβουμε τον σεβασμό ορισμένων ονομάτων ως προϋπόθεση στις εμπορικές συμφωνίες. Το δικό μου ερώτημα είναι Κατά πόσον προσπαθήσαμε να το κάνουμε στα πλαίσια των συμφωνιών οικονομικής συνεργασίας και αν ναι, τι είδους μορφή μπόρεσε να προσλάβει αυτό. Thank you. Um, Maria Η Μαρία Χόιμπρουκ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Λόλε, για την ε, γνωμοδότηση αυτή Πιστεύω πως έχεις καταφέρει να συμπεριλάβεις όλα τα σημεία τα οποία αναφέρουμε και εμείς και αναφέραμε ανέκαθεν να επαναλάβω κι εγώ τη σημασία που έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη σημασία που έχει η τήρηση των ε, μηχανισμών για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών ε, δικαιωμάτων κτλ. Υπάρχουν ορισμένοι τομεί που είναι χαρακτηρισμένοι από ασάφεια στο διεθνέ δίκαιο. Χρειάζεται λοιπόν να ε, αλλάξει αυτό έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και πρέπει φυσικά να συμμετέχουν και οι μεγάλες πολυεθνικέ. Χρειάζεται να αλλάξει η στάση τους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Όχι μόνο όμω οι μεγάλες πολυεθνικέ εταιρείε, αλλά και οι κυβερνήσεις. Δυστυχώ θεωρώ λυπηρό το γεγονός ότι ε, δεν είναι δεσμευτικές ε, οι αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Χρειάζεται λοιπόν η δημιουργία ενός ε, δεσμευτικού οργάνου. Το ανέφερε και ο Σάρλ Γκέρενς ήδη εξάλλου πώς ε, πρέπει να υπάρξει ένα τέτοιο μέσο. η Πολλές φορές οι επιχειρήσεις έχουν την ε, ελευθερία της επιλογής για το αν θα τηρήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή όχι. Αυτό όμως πρέπει να αλλάξει και στην Ευρώπη όμως έχουμε ευθύνη. Πρέπει και εμείς να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι τα εργασιακά πρότυπα. Εδώ πρέπει να τηρηθούν τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και πιστεύω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε επίσης και άλλα ε, πρότυπα. Οι εμπορικές συμφωνίες αναφέρθηκαν ήδη από τους προλελήσαντες. Πιστεύω πως πρέπει να εξετάσουμε ξανά τις εμπορικές συμφωνίες έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει κάποιος μηχανισμός ή κάποιες ρήτρες που να αναφέρονται στον περιβαλλοντικό και στον κοινωνικό παράγοντα. Είναι δική μας η ευθύνη και για την κοινωνία και για το περιβάλλον. Γι' αυτό πρέπει να εργαστούμε προς ε, την προάσπιση των πολιτών και του περιβάλλοντος. Αυτά φυσικά δεν τα λέω για να ασκήσω κριτική στην έκθεση, αλλά για να ε, προτείνω στην εισηγήτρια να συμπεριλάβει τα σημεία λίγο πιο έντονα. Κυρία Χέντι Χαουτάλια, έχετε το λόγο. Ναι, θα είμαι σύντομη δύο σημεία. Καταρχάς πιστεύω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό η Επιτροπή μας να αναλάβει ενεργό ρόλο στην, ε, στο θέμα αυτό με τις επιχειρήσεις, να γίνει διάλογος. Γι' αυτό λοιπόν ε, πιστεύω πως είναι πολύ σημαντική η γνωμοδότηση της ε, κυρίας Σάντζες. Έπειτα πιστεύω πως πρέπει να απαιτήσουμε την εφαρμογή εθνικών ε, σχεδίων που θα ε, αφορούν τις ε, επιχειρήσεις και τα επιχειρηματικά σχέδια και δεν βλέπω κάποια τροπολογία σχετική με αυτό. Είναι ζωτική σημασία οι κατευθυντήριες γραμμές αυτές να εφαρμοστούν. Δεν θέλω βέβαια να προτείνω αντικατάσταση του σημείου 6 της γνωμοδότησης της ε, ΛΟΛΑ που αναφέρεται στις ε, διεθνείς συνθήκες και την ε, διεθνή συνεργασία έτσι ώστε να υπάρξει λογοδοσία για τις ενέργειες των μεγάλων επιχειρήσεων. Η παράγραφος 6 έχει να κάνει με το ότι πολλές χώρες αρνούνται να ε, αλλάξουν τις, ε, τις ε, διατάξεις και να τις κάνουν δεσμευτικές. Και αυτό θέλουμε να αλλάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Φορμεντίνη από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Trade. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, έχετε το λόγο. Πολύ σύντομα παρακαλώ και μετά θα δώσουμε ξανά το λόγο στην κυρία Σάντσες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε τη Digitrade Trade και digit DEFCO και θα θέλαμε να κάνουμε μερικά σύντομα σχόλια. Εισαγωγικά θα ήθελα να πω πόσο με ευχαριστεί το ενδιαφέρον σας για αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο το ενδιαφέρον για θέματα εμπορίου. Ακούσαμε προηγουμένως για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Θα θέλαμε να πούμε ότι προσπαθήσαμε να συνυπολογίσουμε στην ατζέντα του 2030 τη διδάσταση εκείνη που ε, αφορά το εμπόριο. Θα θέλαμε επίσης να αναφερθούμε στις εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην εμπορική πολιτική της Ευρώπης είτε σε μονομερή μέσα, το GSP, GSP+. που συμπεριλαμβάνουν δεσμευτικούς κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εγκαθιδρύουν μια σχέση μεταξύ εμπορικών και πολιτικών συμφωνιών. Το τελευταίο σημείο πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το διεθνές πλαίσιο και τη δουλειά που κάνει αυτή η Επιτροπή. Εμείς αν ανοίξουμε μια ματιά στα ψηφίσματα που υιοθετήθηκαν το 2010, θα διαπιστώσουμε ότι πολλά έχουν αλλάξει στον κόσμο και θα πρέπει να υπάρξει μια διασύνδεση μεταξύ του διεθνούς πλαισίου και της πολιτικής μας. Θα ήθελα να τελειώσω τις παρατηρήσεις μου λέγοντας ότι και στον τομέα του CSR έχουν συμβεί πολλά. Υπάρχουν εργαλεία που δεν υιοθετήθηκαν εκείνη την εποχή, αλλά νομίζω ότι καταβλήθηκε μια προσπάθεια να υπάρχουν κατευθυντήριοι γραμμές για τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να κινηθούν προς την κατεύθυνση της ε, απαιτούμενης ε, προσοχή. Θα ήθελα να δώσω στο συνάδελφό μου, τον Ζωκόκη από την Ζητεύκο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ, εν συντομία, να αναφερθώ σε μερικά μέτρα που θα λείπουν από την υιοθέτηση της σύστασης Παίρνοντα την έμπνευσή μας από το σχέδιο που βρίσκεται μπροστά σας, όπου αναφέρεται ότι θα πρέπει να γίνει μία εκ των προτέρων ανάλυση, θα ήθελα να πω ότι γίνεται μία αξιολόγηση των επιπτώσεων πριν ή κατά τη διάρκεια των εμπορικών διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι κάτι που ενδυναμώθηκε περαιτέρω από την άποψη της πολιτικής συνοχής για την ανάπτυξη. Αυτό είναι μέρος του, του πακέτου για καλύτερη θυσία. Αυτά είναι έγγραφα τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο. Θα ήθελα εν συντομία να αναφερθώ τη δουλειά που έχει γίνει σε διαφάνεια σε συγκεκριμένους ε, ε, τομείς. Ε, μερικές ε, από τις οδηγίες μας πρόσφατα τροποποιήθηκαν για να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά την δραστηριότητα των διεθνών εταιριών οδηγία, η στρατηγική για την εταιρική ευθύνη επαναπροσδιορίζεται εδώ και δίχως άλλο θα επαναξεταστούν όλα τα στοιχεία που αναφέραμε εδώ. Και αυτή θα είναι μια επιπλέον ευθύνη για το Κοινοβούλιο να συνεισφέρει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχει ναι, σύντομα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκεί πίεση στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να αλλάξει κάτι στις ε, κατευθύνες γραμμές ράγκη. Maybe you have to, if, you, Εάν δεν γνωρίζετε, μπορείτε να απαντήσετε αργότερα. Δεν σας άκουσα καλά και εγώ τι, πώς, πώς είπατε. είναι οι αρχές ε, ράγκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιέσει τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να πιέσουν και εκείνα για την εφαρμογή τους. Θέλω να τους ε, ρωτήσω λοιπόν. Ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανέλθει με την απάντησή της σε αυτή την Επιτροπή. Η κυρία Σάντσες. Σας ευχαριστώ Λίντα. Θα είμαι πολύ σύντομη. Όμως θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Θέλω να πω για την πραγματικότητα για την θέση για την οποία έκανε λόγο ο συνάδελφος για αυτήν την γνωμοδότηση είναι η πραγματικότητα όμως. Εμείς αντανακλούμε στο έγγραφο την πραγματικότητα εκτός των συνόρων μας και πολλοί υφίστανται τα πάνδυνα. Δεν είμαστε εχθροί του εμπορίου, ούτε εχθροί των επιχειρήσεων. Είμαστε εχθροί εναντίον εκείνων που παραβιάζουν τα δικαιώματα του ανθρώπου όπου και να τα παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο. Έχουμε εμπορικές καταστάσεις που είναι τρομακτικές με μεγάλες ε, επιχειρήσεις που δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Ούτε υπάρχουν κυρώσεις εις βάρος τους, ούτε υπάρχει λογοδότηση. Και είναι πολλές επιχειρήσεις και ισπανικές κλωστοϊφαντουργικών που υπάρχει μια μικρή ελάχιστη τυποτένια αποζημίωση το πολύ πολύ που επιδικάζεται και δεν μπορεί κάτι τέτοιο να ισχύει. Εμείς δεν θέλουμε να παραβιάζονται τα δικαιώματα. Το εμπόριο είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο για την ανάπτυξη και όχι ως τροχοπέδι φρένο για την ανάπτυξη. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε και πρέπει να διευρύνονται τα δικαιώματα. Τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν είναι επαναστατική πράξη. Υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι αυτό συμβαίνει. Όμως εμείς μας αντιμετωπίζουν ως επαναστάτες επειδή ζητάμε να είναι σεβαστά τα δικαιώματα του ανθρώπου. Είναι το εμπόριο και επιχειρήσεις όμως που πρέπει εκείνοι και εκείνες να ε, προσαρμοστούν στα δικαιώματα του ανθρώπου και όχι αντίστροφα. Και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχόλιο όταν ήμουν στη Γενέβη <clears throat> κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτής της Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για μια δεσμευτική συμφωνία ώστε οι πολιεθνικές να σέβονται τα δικαιώματα του ανθρώπου εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλο το πρωί προσπάθησε να τροχοπεδίσει επανειλημμένα την ε, δημιουργία μιας τέτοιας συμφωνίας. Ήταν η πίεση των πολιτών εκείνη τη στιγμή, όλοι άσκησαν πίεση και δεν ήθελαν να υπάρξει μια τέτοια πιστοδρόμηση. Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν τρομερή, τρομακτική κατάσταση και η θέση της για αυτό το θέμα. Και ο αποκαλούμενος εκπρόσωπός της προσπάθησε να τροχοπεδίσει τα πράγματα επανειλημμένα ώστε να μην προχωρήσει μια τέτοια συνθήκη, μια τέτοια συμφωνία. Και για να ολοκληρώσω θα πω ότι συμφωνώ με αυτά που έλεγε η Λίντα κάνουμε λόγο για συστάσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη από το 2010, αλλά πρέπει να είναι πιο αυστηρές, πιο δεσμευτικές, ε, ώστε να είμαστε σε θέση πραγματικά να είμαστε πιο στεναροί και αποτελεσματικοί για αυτό το θέμα, που έχει σημασία ε, κλειδιού για πάρα πολλούς ανθρώπους παγκόσμια. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τη συνεργασία σας και την κατανόηση. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες 23 Σεπτεμβρίου. Αύριο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, συνάδελφοι. Μην αργήσετε, μην μακρηγορήσετε, να συγκεντρωθείτε στην ουσία. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για αυτό το θέμα. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο. Ε, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας, κύριε, κυρία Διευθύντρια της ε, Δείξα Δείξατε μεγάλη υπομονή, μας περιμένατε 15 λεπτά μέχρι να τελειώσουμε τα προηγούμενα σημεία. Έχουμε χρόνο. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που καταφέρατε να έρθετε. Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στην Επιτροπή μας και εύχομαι να έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία τα επόμενα χρόνια. Φυσικά είναι δύσκολες οι εποχές. Χθε συζητήσαμε με τον Επίτροπο Μίμητσα και αναφέρθηκε στο καταπίστευμα για την Αφρική που θα ιδρύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι γίνονται κάποιες συζητήσεις στο Συμβούλιο έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που έχουν προκύψει με την, από την εισρωή των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ιδιαίτερα σημαντική έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την κρίση των προσφύγων και να τους στηρίξουμε στην γειτονία μας. Και ο λόγος για τον οποίο ζήτησα να συζητήσουμε το θέμα αυτό σήμερα είναι ότι οι πολίτες μας ρωτάνε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ακούμε ότι ε, διακόπτεται η επιστημιστική βοήθεια στην Ιορδανία και τον Λίβανο. Ε, ακούμε ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Αληθεύει ότι τα κονδύλια συγκεντρώνονται αλλά μετά δεν προχωρούν. Είναι Μία πολύ σημαντική συζήτηση πιστεύω. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και είναι πολύ χρήσιμο να συζητήσουμε, να δούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι περισσότερο πρέπει να κάνει έτσι ώστε η ανθρωπιστική βοήθεια να παρέχεται με έναν τρόπο που είναι σωστός. Κυρία Γενική Διευθύντρια, θα σας δώσω το λόγο για περίπου 10-15 λεπτά και μετά θα ακούσουμε τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όπως σας είπε η κυρία Πρόεδρος ανέλαβα την 1η Σεπτεμβρίου και ένα από τα πρώτα μου καθήκοντα ήταν να συναντήσω την πρόοδό σας. Εγώ ήθελα να σας δω νωρίτερα, αλλά Συνέβησαν πολλά και δεν ε, μπόρεσε να γίνει η συζήτηση όταν ήθελα. Έχω μαζί μου τον Ελπίδη Φένα. Παρακαλώ, εάν έχετε κάτι να πείτε, σας παρακαλώ, εκτός της αίθουσας. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορώ να, να ακούσω από εδώ τα όσα λέτε μιλώντα. Είναι δύσκολο λοιπόν η κυρία να συγκεντρωθεί. Ε, ενδεχομένως υπάρχουν ε, ερωτήσεις που θα θέλετε να κάνετε και οι συναδελφοί μου θα μπορέσουν να σας δώσουν απαντήσεις σε περίπτωση δεν ξέρω εγώ. Όπως σας είπα, αυτή η κρίση με τους πρόσφυγες είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις με την οποία βρέθηκε αντιμέτωπη η Ευρώπη. Πιστεύω ότι τα όσα είπε πρόσφατα ο κύριος Γιούνκερ δείχνουν τη σοβαρότητα της ε, κρίσης. Είναι σαφές ότι η Επιτροπή, όπως και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και οι χώρες μέλη κατανοούν το πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα και πόσο αναγκαίο είναι να δοθεί η κατάλληλη απάντηση σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε αυτό που γίνεται στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Επιτροπής ήθελε να σας μιλήσει για αυτό το θέμα. Σε επίπεδο επιτροπής είναι και για μας μια στιγμή για να προσπαθήσουμε να υπάρξουν οι περισσότερες συνέργειες μεταξύ των διαφόρων μηχανισμών που έχουμε για να απαντήσουμε σε αυτή την κρίση που έγινε μια εσωτερική κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά που έχει τις ρίζες της έξω. Μια κρίση και για τις χώρες προέλευσης αλλά και τις χώρες διέλευσης που βρίσκονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών που αντιμετωπίζουν μια βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάθεση. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε απόλυτη συνείδηση αυτού και ότι συνεργαζόμαστε με τις διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής. Συνεργαζόμαστε με τη Γενική Διεύθυνση διεύρυνσης με τη διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων, έτσι ώστε να υπάρξει μια όσο γίνεται καλύτερη συνεργασία. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα. Καταρχάς, σε αυτό που κάνουμε εμείς σε Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας, σε ό,τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σε επίπεδο εσωτερικό και εξωτερικό. Σε επίπεδο εσωτερικό, πέρα από αυτή τη στενή συνεργασία με τους συναδέλφους, θα πρέπει να έχουμε την βεβαιότητα ότι υπάρχει συνέργεια μεταξύ των διαφόρων τομέων σε επίπεδο πολιτικής, γετνίας ή διάφορα μέσα για την ανάπτυξη. Διεξάγεται και μία συζήτηση από τον Ιούλιο για να υπάρξουν όσο κινείται περισσότερες συνέργειες για να υπάρξει ελαστικότητα μεταξύ των διαφόρων μέσων του προϋπολογισμού γνωρίζοντας ότι υπάρχει περισσότερη ελαστικότητα από ό,τι άλλες γενικές διευθύνσεις στη διαχείριση των πιστώσεων. Ένα άλλο μέσο είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Πολιτική Προστασία. Ξέρω ότι μερικοί από εσά έγραψαν στον Επίτροπο Στυλιανίδη για να ζητήσουν να ενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός. Σας απάντησαν, αλλά είναι μία ευκαιρία για να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα. Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να δραστηριοποιηθεί, να τεθεί σε εφαρμογή μόνον κατόπιν αιτήματο μιας χώρας που συμμετέχει. Δηλαδή η ίδια η Επιτροπή δεν μπορεί να ενεργοποιήσει η ίδια αυτό το μηχανισμό. Εμείς δηλαδή ως Επιτροπή δεν μπορούμε να τον θέσουμε σε εφαρμογή ακόμα και κατόπιν αιτήματό σα. Αυτή η ενεργοποίηση θα πρέπει να γίνει από ένα από τα συμβαλόμενα μέρη. Αυτό συνέβη και με την Ουγγαρία, η οποία έθεσε σε εφαρμογή πριν από μερικές μέρες αυτό το μηχανισμό, επικαλούμενη την ε, αλληλεγγύη των άλλων χωρών που συμμετέχουν έτσι ώστε να, αποκτεί, να, έχει πρόσβαση σε αυτά που είχε ανάγκη για να μπορέσουν να ε, αντιμετωπίσουν αυτό το κύμα προσφύγων. Το ίδιο και με τη Σερβία, δραστηριοποίηση, ενεργοποίηση μηχανισμού για να υπάρξει συμμετοχή των άλλων συμβαλωμένων μερών για να υπάρχει παροχή αυτοκινήτων, καυσίμων, οχημάτων, καυσίμων κτλ. Από ε, αυτός ο μηχανισμός έχει τεθεί σε εφαρμογή. Αν η Ελλάδα, η Ιταλία επιθυμούν να θέσουν σε εφαρμογή αυτό το μηχανισμό, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες έτσι ώστε να υπάρξει ανταπόκριση στις ανάγκες τους. Αλλά μέχρι στιγμής ούτε η Ελλάδα ούτε η Ιταλία δεν ενεργοποίησαν αυτό το μηχανισμό. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο που θα πρέπει να υπογραμμίσουμε γιατί υπάρχει κάποια παρανόηση σχετικά με το θέμα της ενεργοποίησης του μηχανισμού. Το κατά, το κατά πόσο δηλαδή μπορεί κανείς να το χρησιμοποιεί όσο ε, συχνά θέλει. Αύριο θα πάω στο Λουξεμβούργο, θα γίνει μια ε, διεύθυνση με τους γενικούς διευθυντές πολιτικής προστασίας των μελών του μηχανισμού. Θα είναι μια ευκαιρία για μένα να ευαισθητοποιήσω και πάλι αυτές τις χώρες και να συμβάλλουν στην ενεργοποίησή του ότι αυτός ο μηχανισμός βρίσκεται εκεί για να υπάρξει ελληνική μεταξύ το κορώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βοηθηθούν οι χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε ό,τι αφορά αυτό το ρεύμα προσφύγων. Η δράση της Ένωσης είναι άλλης φύσης. Εκεί παρεμβαίνουμε για μια οικονομική βοήθεια στις διεθνείς οργανώσεις, στις ε, ΜΚΟ και στις οργανώσεις μέλη των Ηνωμένων Εθνών, που είναι οι πρώτοι συνομιλητές σε επίπεδο ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά την φύση της κρίσης πέρα από την μεταναστευτική κρίση που είναι ο μηχανισμός που πυροδοτεί τα όσα συμβαίνουν τώρα, είναι σαφές ότι πρόκειται για μια κρίση προσφύγων. Και η κρίση στη Συρία είναι αυτό που το καθοριστικό στοιχείο. Εκατομμύρια Σύριοι οι οποίοι εγκαταλείπουν τη Συρία χωρίς να υπολογίσουμε τα εκατομμύρια των εκτοπισμένων στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό το κύμα προσφύγων θα συνεχίσει να έρχεται στην Ευρώπη στο βαθμό που δεν έχει ρυθμιστεί το πρόβλημα στη Συρία. Είναι σαφές ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει μια γενικότερη λύση και πιστεύω ότι ένα από τα μηνύματα του Προέδρου Γιούνκερ στην ομιλία του ήταν ακριβώς αυτό. Η Ευρώπη είναι ένας από τους βασικούς δωρητές εδώ. Θα ήθελα να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τις Ηνωμένε Πολιτείες παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η Ένωση μέχρι στιγμής έχει συμβάλει με 4 δισεκατομμύρια ευρώ 4 δισεκατομμύρια λοιπόν ευρώ για την κρίση στη Συρία από την αρχή και το 1, εκατομμύριο, 1 δισεκατομμύριο ήταν για ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά είναι σαφές βεβαίως ότι υπάρχει ένα έλλειμμα χρηματοδότησης. Από αυτή την άποψη οι εκκλήσεις των ε, Ηνωμένων Εθνών καθιστούν σαφές ότι οι εκκλήσεις αυτές καλύφθηκαν κατά 30% και αυτό αυτό οδήγησε σε μία περικοπή της βοήθειας από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε, να, να απελευθερώσουμε επιπρόσθετα κονδύλια. Αυτό είναι κάτι που θα παρουσιάσουμε αύριο στα στην ε, Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής. Θα δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσουμε θα μπορέσουν να υπάρξουν επιπρόσθετα κονδύλια για να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές που καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτό το κύμα προσφύγων, την Τουρκία, τη Σερβία, την, ε, το Φύρομ Θα ήθελα επίσης να θυμίσω ότι επικεντρωνόμαστε στην κρίση στη Συρία για απόλυτα αιτιολογημένους λόγους. Θα ήθελα να θυμίσω ότι ο οδός των Βαλκανίων δεν είναι η μοναδική οδός από την οποία σειραίουν πρόσφυγες, θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε και σε άλλες κρίσεις, στη Λιβύη για ε, παράδειγμα που είναι ένα άλλο σημείο από όπου προέρχονται μεταναστευτικά καρέματα προς την Ευρώπη. Δεν θα ήθελα να μιλήσω περαιτέρω για τα προβλήματα στην Ιεμένη ή σε άλλα μέρη του κόσμου που υπάρχουν σημαντικές μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρισκόμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με μια ε, μείζωνα κρίση και θα πρέπει να δοθούν πολιτικές και όχι μόνο ανθρωπιστικές απαντήσεις. Η ανθρωπιστική απάντηση είναι η πρώτη βεβαίως που θα πρέπει να δοθεί. Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί σε επίπεδο επιτροπής για να ε, αυξηθεί η ενίσχυση που μπορούσαμε να δίνουμε. Ε, αυτά ήθελα να πω. Βεβαίως είμαι στην διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες. Θα ήθελα όπως να περιοριστώ εδώ για να σας δώσω τη δυνατότητα να πάρετε και εσείς το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και μας παρουσιάσατε αυτές τις πληροφορίες και μας είπατε αυτά που μπορεί και δεν μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο εσωτερικό τη Θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη, στα πλαίσια διάσκεψη την ανθρωπιστική βοήθεια, όπου θα συζητηθεί το πόσο πρέπει να είναι αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά πολλοί μας λένε ότι δεν τα πάμε καλά εντός των συνόρων μας. Πώς θα γίνει να, να βοηθήσουμε εκτός των συνόρων μας. Πολλοί μας ρωτάνε, μα, μα τι γίνεται επιτέλους ιδιαίτερα μάλιστα στα σύνορα, στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Ο Ενρίκε Γκερέρο θα πάρει το λόγο πρώτος, ο οποίος έχει αναλάβει και την έκθεση για την ανθρωπιστική βοήθεια και μετά ο Νταβοστίερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρότι είχα την ευκαιρία να συνέλθω αμέσως μετά από τον διορισμό σας να συναντηθούμε. Είναι καλό νομίζω αυτό το οποίο γίνεται. Διότι όπως είδαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις τελευταίες εβδομάδες, στις Ολομέλειες για παράδειγμα, υπάρχουν δύο εμπλεκόμενοι που συμμερίζονται τη διάγνωση και την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα προβλήματα και λύσεις που είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η μεγάλη πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου και υπάρχει και άλλος εμπλεκόμενος, τα κράτη-μέλη στο σύνολό τους, στο Συμβούλιο, πως τόσο πόρο απέχουν από αυτή τη συμφωνία να δράσουμε, να δράσουμε γοργά κιόλα και να δράσουμε με αποτελεσματικό τρόπο. Και γι' αυτό πιστεύω ότι σήμερα για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθυγραμμίζονται, βρίσκονται στην ίδια πορεία. Πρέπει αμέσως να αναφέρω <clears throat> με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και ερωτήματα. Πρωτού κάνω τις συγκεκριμένες ερωτήσεις, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Η πρώτη, Όλοι θα θυμούνται ότι την πρώτη απόφαση, την πρώτη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έγινε για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση των προσφύγων και μεταναστών ή των ετούντων άσυλο τέλος πάντων έγινε το Μάιο. Σήμερα ουσιαστικά φτάνουμε στο μήνα Οκτώβριο, δηλαδή πέρασαν πέντε μήνες, τέσσερις μήνες και κάτι και μόνο την προηγούμενη εβδομάδα ή δύο εβδομάδες πριν <clears throat> φτάσαμε σε μια συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών ώστε να υπάρξει ανακατανομή των 40.000 που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατανεμηθούν κατά το Μάιο. Ωστόσο, εντωμεταξύ η διάσταση προφανώς των ροών αυτών προσφύγων και μεταναστών έχει αυξηθεί γεωμετρικά και σε σχέση με τις ε, δράσεις ε, από το προηγούμενο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και που δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τους 120.000 σε σχέση με παράδειγμα που θα έπρεπε να φύγουν αυτοί από την Ιταλία, την ε, Ελλάδα και την Ουγγαρία και να κατανεμηθούν ε, ισομερώς ε, στα κράτη-μέλη. Έχουμε λοιπόν το μεταξύ εκατοντάδες χιλιάδες άτομα που περιπλανώνται σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και αναζητούν ασφαλές κατάλημα. Πέρασαν τέσσερις μήνες χωρίς να βρεθεί μια λύση που να είναι βιώσιμη και εφαρμόσιμη άμεσα από πλευρά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται λοιπόν. Εν τω μεταξύ πρέπει να επισημάνουμε φυσικά ότι οι πολίτες, η κοινωνία των πολιτών, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δράσανε, έδρασαν άμεσα επί τόπου και ανακούφισαν τουλάχιστον εν μέρη μερικώς τις ανάγκες και τα δεινά που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι. Τους ανακούφισαν. Αν δούμε τώρα αυτό το οποίο τίθεται από τη Γενική Διευθύντρια και που βρίσκεται στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτά τα μέσα αυτά τα μέσα μπορούμε να τα ενεργοποιήσουμε αλλά προφανώς αυτά τα μέσα δεν είναι ικανά να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση στη διάσταση που έχει των τόσων πολλών προσφύγων και γι' αυτό χρειάζονται δεσμεύσεις, δεσμεύσεις των κρατών μελών, πολύ παραπάνω από αυτές τις δεσμεύσεις που μπορούν να επιτευχθούν μέσω της Επιτροπής με τα μέσα που έχει. Και πρέπει να υπογραμμίσουμε, χωρίς να επεκταθώ περισσότερο σε αυτό, ότι αυτή η κρίση δεν είναι μόνο μια σημαντικότατη κρίση για τις διαστάσεις που έχει, διότι έχει επιπτώσει στα άτομα, εκατοντάδες χιλιάδες που την υφίστανται, αλλά είναι μια κρίση για την Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί σε κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι μόνο σε κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε κρίση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι λοιπόν η χρονική στιγμή να δράσουμε και να εκφραστούμε. Το κάναμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα εμείς με μια στεναρή διαζώσης φωνή να υψώσουμε τη διαμαρτυρία μας έναντι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί αύριο από τους Υπουργούς ώστε να καταλήξουν σε μια συμφωνία ώστε να μπορέσουν να ανακουφιστούν αυτά τα άτομα που υφίστανε τα πάνδυνα. Εδώ και δύο εβδομάδες είχαμε μια εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχαμε και την παρουσία του είπα του εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες του κυρίου Γκουτέρες Πορτογάλου και της κυρίας Φεντερίκα Μοντερίνη και του κυρίου Αβραμόπουλου και ήταν σαφές σε αυτή την εκδήλωση ότι ταυτόχρονα ενώ προσπαθούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα μέσω πρόθεσμα πρέπει άμεσα να δράσουμε. Αυτό είναι το πιο αναγκαίο. Να δράσουμε άμεσα, πρόθεσμα αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες και τα δεινά αυτών των ανθρώπων. Περνάω στις ερωτήσεις, σε μια αξιολόγηση που θα ήθελα να μας δώσει, αν την έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όποια και να είναι η προέλευση αυτών των κονδυλίων, τα ποσά των κονδυλίων αυτών. Για ποια κονδύλια μπορεί να γίνει λόγος για τα οποία θα χρειαζόμαστε για να καλύψουμε επαρκώς ε, τις ανάγκες αυτής της κρίσης προσφύγων που έχουμε. Και τι κάνει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξει τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις <clears throat> που δρούν επιτόπου στις διάφορες χώρες και που έχουν μεγάλα κενά χρηματοδότησης και πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες χρηματοδότησής τους για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και των άλλων οργανώσεων που τοπικά δραστηριοποιούνται στη Λιβύη, η Ορδανία και αλλού για παράδειγμα. Και είναι αυτονόητο φυσικό και λέω ότι η διευθύντρια της ΕΚΟ θα συμμερίζεται αυτή την ιδέα μου ότι δεν μπορεί να επιληθεί απλά και μόνο με μια προοπτική ασφάλεια σε αυτή η κρίση πρέπει να επιληθεί με μια επικέντρωση ανθρωπιστική, ανθρωπιστικής βοήθειας. Πρέπει στο Συμβούλιο αύριο να ληφθεί υπόψη αυτό. Δεν είναι μόνο το πώς θα διαφυλάξουμε σύνορα και πώς θα δώσουμε κονδύλια για να διασφαλίσουμε την εξωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε εκείνους που βρίσκονται εντός και εκείνους που θα μπορέσουν να φτάσουν ίσως ώστε με τον πιο ασφαλή τρόπο να δημιουργήσουμε διαδρόμους ανθρωπιστικούς να μπορούν ε, να αντιμετωπιστούν τα προβλήματά τους. Θέλω να αναφέρω μια φράση που αναφέρθηκε ήδη και όχι μόνο από μένα αλλά από πολλούς άλλους φυσικά αλλά νομίζω συνθέτει με πολύ καλό τρόπο το πρόβλημα που έχουμε. Είναι μια φράση που είπε ο Γιούγκερ για την κατάσταση της Ένωσης που είπε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα δύο αυτά που σε αυτή την κρίση. Το τονίζω. Αν δεν θέλουμε λοιπόν να μειωθεί η Ευρώπη, λιγότερη Ευρώπη και λιγότερη Ένωση, αύριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δράσει με αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Στήρ και η κυρία Μπεσέρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τη Γενική Διευθύντρια. Και εμείς θέλουμε από την πλευρά μας να πούμε ότι χρειάζεται μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτήν την ε, κρίση των προσφύγων. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε να παρατηρούμε αυξανόμενες εντάσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη το είδα στην Κροατία να συμβαίνει αυτό, στην πατρίδα μου. Είδα τις ε, εντάσεις στα σύνορα με την Σλοβενία, για παράδειγμα, το περασμένο Σαββατοκύριακο. Καθώς επίσης και το τι γίνεται στα σύνορα Κροατίας και Ουγγαρίας, μετά στα σύνορα Ουγγαρίας-Σερβίας. Υπάρχουν ε, μέτρα, αντιδράσεις αυτά τα μέτρα και μετά βλέπουμε ένα εναντίον ενός, δύο εναντίον τριών και ούτω καθεξής. Αυξάνονται λοιπόν οι εντάσεις, γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, εάν δεν θέλουμε να δούμε όχι μόνο να αυξάνονται οι εντάσεις, αλλά να οδηγούμαστε και σε σειράξεις στα σύνορά μας, το οποίο είναι φυσικά κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί πριν από λίγα ε, χρόνια. Τώρα κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Αναφερθήκατε στην βοήθεια στη Σερβία, τη Μακεδονία. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι είδους βοήθεια είναι αυτή. Ε, θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν πιο ασφαλή διάδρομο διέλευσης ή να φροντίσουμε τους πρόσφυγες μέσα σε αυτές τις χώρες. Είναι σημαντικό να δούμε ποια είναι η προσέγγιση ε, δική σας για την βοήθεια αυτή. Επίσης, μια παρόμοια ερώτηση έχω για την Τουρκία, όπου φυσικά υπάρχουν δύο εκατομμύρια πρόσφυγες. Πώς εξελίσσεται ο διάλογος με τις τουρκικές αρχές. Διότι η Τουρκία είναι από τις ε, χώρες όπου από πού πηγάζουν αυτές οι ροές. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικός, ουσιώδης θα έλεγα, ο διάλογος με την Τουρκία. Όχι μόνο ε, χρειάζεται οικονομική υποστήριξη, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι στάση τηρούν οι αρχές στην Τουρκία. Ευχαριστώ πολύ, Μπέτριξ Πεθέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Γενική Διευθυντή για την σαφέστατη τοποθέτηση σε σχέση με τη δράση από πλευράς υπηρεσίας ΕΚΟ Συμφωνώ απόλυτα με τον Ενρίκε. Χαίρομαι που ανέφερε πολλά από αυτά που ήθελα να πω και έτσι δεν θα επιμείνω περισσότερο σε αυτά. Πιστεύω οπωσδήποτε ότι είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι η ανθρωπιστική απάντηση χορηγείται κατά πρώτη γραμμή και είναι εκείνη που πρέπει να διασφαλιστεί πρώτη. Αλλά μέσω της πολιτικής μας των θεσμικών οργάνων φαίνεται ότι υπάρχουν μόνο δύο θεσμικά όργανα που έχουν ε, γνωρίσει, που έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη αυτής της πολιτικής και πρέπει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού να το συνειδητοποιήσει για να δράσει. Αυτό το οποίο καταδεικνύεται μεταξύ άλλων είναι η ανικανότητα των κρατών να δουν λίγο πιο πέρα από τα κοντόθωρα ε, μειοπικά εθνικά τους ε, συμφέροντα και να δουν την εικόνα και τις ανάγκες σφαιρικότερα και στην ε, Ισπανία και την κατάσταση δεν υπάρχει η ικανότητα να δοθεί απάντηση αποτελεσματική και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να τονίσουμε ότι τα κράτη σε αυτές τις προόδους, σε αυτές τις προβλέψεις για κονδύλια που θα στοχεύσουν για τους πρόσφυγες που τελικά θα καταλήξουν στη χώρα τους, δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα κονδύλια αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται απλώς λόγος για κονδύλια και βρισκόμαστε σε εκλογική περίοδο όπως στην Ισπανία και αυτό είναι ένα μέσο ε, εκλογικής, ας το πω έτσι, εκλογικών ελιγμών. Κάτι το απαράδεκτο, το αναξιοπρεπές. Και πέρα από αυτό για την αξιολόγηση που εσείς κάνετε για το ποιες είναι οι ανάγκες για κονδύλια που θα χρειαστούν όχι μόνο για να δώσουμε επαρκή προσοχή στις ανάγκες αυτού, του αριθμού προσφύγων όταν γίνεται λόγος για 120.000 που θα μετεγκατασταθούν ποια είναι η πραγματική αξιολόγηση για αυτούς τους ανθρώπους στους οποίους θα πρέπει να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια που βρίσκονται ήδη στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα καταλήξουν, θα φτάσουν σε αυτήν ώστε να διασφαλίσουμε ότι όχι μόνο θα γίνουν δεκτά αυτά τα κονδύλια αλλά να δούμε πώς αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια που έχει θα πρέπει να έχει μια διάρκεια, διότι δεν πρόκειται μόνο για την άφηξη ή την αναχώρηση αυτών των ατόμων, για τη διάρκεια εγκατάστασής τους πώς αυτός ο μηχανισμός θα μπορέσει να ενεργοποιηθεί ώστε να λειτουργήσει και να παράσχει αυτά τα κονδύλια. Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση έχω και θα ήθελα στον προλαλήσαντα και στην ερώτησή του να προσθέσω αυτήν. Πώς δηλαδή μπορούμε να βοηθήσουμε και από την άλλη πλευρά πώς μπορείτε να υπομισθείτε την ευθύνη πώς μπορεί να υπάρξει προθυμία να υπομισθούν οι υπεύθυνοι αυτοί, αυτές τις ευθύνες και δεν μπορώ να φανταστώ ποιος μηχανισμός είναι εκείνος που θα μπορέσει όλα αυτά να τα καλύψει αποτελεσματικά στην αναζήτηση αυτής της λύσης που θα πρέπει όλοι να συμμετάσχουν. Πώς το συζητάτε εσείς από δική σας πλευράς, γιατί κάνουμε λόγο για την Ευρώπη μας, για μια ένωση αξιών που είναι η Ευρώπη, αλλά πρέπει από την άλλη πλευρά να δούμε με τα προβλήματα αν αφαιθούν κάποιοι μόνοι τους Πρέπει να δούμε πώς θα υπάρχει η προθυμία οικονομικά ή και πολιτικά να υπάρξει συμμετοχή ώστε να του ανακουφίσουμε. Τι προβλέπετε, τι σκέπτεστε εσείς ώστε όλα αυτά να μπορέσουν να καλυφθούν επαρκώς. Διευτεμέρα παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είσαστε πολύ νέοι όλοι σας. Εγώ είμαι λίγο πιο ηλικιωμένος και θέλω να υπενθυμίσω σε σας κάτι κάποια παρόμοια γεγονότα στην Επιτροπή Μεταναστών ε, σε σχέση με το Συμβούλιο της Ευρώπης είχα συμμετάσχει όσον αφορά τα προβλήματα αυτά των τελευταίων Βαλκανικών πολέμων και είχα την ευκαιρία να δω στρατόπεδα προσφύγων <clears throat> Στάνκοβιτς 1 και το Στάνκοβιτς 2 στην Μακεδονία και το τι γινόταν σε σχέση με, αυτές τις, ε, ε, ε, με αυτή την κατάσταση. Ήταν πολύ δραματική αυτή η ιστορία της πρόσφατης ιστορίας της Ευρώπης και των σειράξεων που είχαν συγκλονίσει την Ευρώπη και στο ανθρωπιστικό επίπεδο. Να μην ξεχνάμε και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό ότι το σημείο 22 στην ημερήσια διάταξή μας λέει ανθρωπιστική απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρίση των προσφύγων. Δεν κάνουμε λόγο για ασφάλεια σύνορων, αλλά μόνο για ανθρωπιστική διάσταση αυτού του προβλήματος. Να το λάβουμε υπόψη. Ακολουθώ το μύτο της Αριάννης στην προηγούμενη συνέχεια επιχειρημάτων για το τι πρέπει να γίνει. Η Γερμανία ήταν επίσης η πρώτη που έδωσε αυτή την απάντηση και πήρε εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα προβλήματα γνωρίζοντας το τι έπρεπε να κάνουν και το κάνουν σε σχέση με την ε, ε, υποδοχή αυτών των ε, ανθρώπων. Τώρα, τα κονδύλια, ο μηχανισμός, πώς μπορεί να δρομολογηθεί και, τα, και οι μηχανισμοί, οι δημοσιονομικοί, πρέπει να μπορέσουν να λειτουργήσουν όχι για να αντιμετωπιστεί το κατεπήγον μόνο, αλλά η ανάγκη αυτή που είναι έκδηλη, ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Το είπε ο Αντώνιο Γουτέρες πρόσφατα, ότι Κονδύλια, κονδύλια, κονδύλια πρέπει να διατίθενται, να διατεθούν. Και αυτό πρέπει να γίνει. Λεφτά, χρήματα χρειάζονται. Και πρέπει λοιπόν για αυτές τις δράσεις ε, με την μεγάλη πείρα που έχουν στην αντιμετώπιση της ε, άμεσης βοήθειας που πρέπει να δίνεται πρωτογενός και δευτερογενός στους πρόσφυγες να δράσουμε. Αν συμφωνείτε λοιπόν πραγματικά για το πρόγραμμα του Μαΐου της ανακατανομής προσφύγων στο οποίο έγινε αναφορά η επανεγκατάσταση όχι μόνο η επανεγκατάσταση των 20.000 των πρώτων ε, των 120.000 Τώρα δεσμευόμαστε για την ε, εποπτεία του κυρίου Γκουτέρες ε, υπό τη δική του εποπτεία του ΙΠΑ του εκπροσώπου των Ηνωμένων για τους πρόσφυγες θα έπρεπε να λειτουργήσει αυτή η δράση. Τώρα, σε σχέση με την συνάδελφο ε, πρέπει να πω ότι η άγνοια είναι πολύ συμβατή με την τόλμη, με την τολμηρότητα. Και η αναφορά που έγινε για την Ισπανία είναι υποδειγματικό παράδειγμα πρόληψης ε, και προληπτικής δράσης. Και πρέπει εδώ να προσθέσουμε για αυτούς που δεν το γνωρίζουν ότι τα κονδύλια που δέσμευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πρόσφυγες, λόγια δηλαδή τα οποία πάλι από τον κύριο Γιούγκερ αναφέρθηκαν 6.000 ευρώ είναι για κάθε ένα από τους πρόσφυγες και απορρέουν από τη δράση επανεγκατάστασης. Αλλά όπως λέω δεν είναι θέμα αυτή τη στιγμή αυτό. Εκείνο όμως θέλω, που θέλω να κάνω είναι να ρωτήσω κάτι τη Γενική Διευθύντρια όσον αφορά την δραστηριοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Λοιπόν, να το δούμε αυτό, γιατί δεν το κατανοώ και δεν το κατανόησα. Δεν το ζήτησαν, λέει, ούτε η Ελλάδα ούτε η Ιταλία να δραστηριοποιηθεί, να δρομολογηθεί. Μυστηριώδες αυτό, πραγματικά κατανόητο. Δεν μπορώ να το συλλάβω και να το κατανοήσω. Πείτε μας, κυρία, σας παρακαλώ πολύ, ποια είναι τα μέσα τα χρηματοοικονομικά μέσα για να καλυφθούν οι ανάγκες της άμεσης δράσης ανθρωπιστικά. Εμένα δεν ε, είναι σημαντικό να μου πείτε υπάρχουν 4 δισεκατομμύρια εκ των οποίων ένα δις θα δοθεί για την ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν είναι αυτό το οποίο είναι το ε, αποτελεσματικό. Όπως λέει ο Αντώνιο Γκουτέρες αυτό είναι απόλυτα ανεπαρκές και λέμε ότι είμαστε οι πρώτοι που δρούμε παγκόσμια και που παρέχουμε αυτή τη βοήθεια και κοιτάξτε πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, αναμένω την απάντησή σας. Ευχαριστώ. Okay, thank you. Um, σας ευχαριστώ πολύ. Για τη Χάουταλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στη συζήτηση που είχαμε σήμερα το πρωί όπου συζητήσαμε το πρόβλημα της ε, ανθρωπιστικής βοήθειας και το ότι εκείνη δεν φτάνει στο στόχο της. Θα ήθελα να ρωτήσω την Γενική Διευθύντρια. Παρακαλώ, μπορείτε να με ακούσετε, γιατί έχω μία ερώτηση απευθείας σε εσάς. Ναι, ναι, δεν μπορούσε να διαβάσει το όνομά σας. Εντάξει, λύθηκε το πρόβλημα. Επανέρχομαι λοιπόν. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν φτάνει τον στόχο της στην Ανατολική Ουκρανία. Πολλοί οργανισμοί εκφράζουν ανησυχίες για το ότι το Κίεβο, για λόγους εσωτερικής ασφάλειας, δεν επιτρέπει στην ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει σε περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας, οι οποίες ελέγχονται από αντάρτες. Και αυτό φυσικά δυσχεραίνει την ε, κατάσταση στην οποία ζουν οι κάτοικοι εκεί, οι πολίτες και δυσχεραίνει και την επικοινωνία ανάμεσα στο Κίεβο και τις περιοχές όπου υπάρχουν αντάρτες. Μία από αυτές τις ε, περιοχές, ε, εκτός Ουκρανίας τώρα, είναι ένα στρατόπεδο έξω από την ε, Δαμασκό, το οποίο ελέγχει το Ισλαμικό κράτος. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ, ο Σαρλ Γκάρεντς. Κυρία Πρόεδρε, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ότι οι χώρες μέλη γενικά δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων, είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να πούμε. Ο προϋπολογισμός που θα ψηφιστεί για του χρόνου είναι, έχει λιγότερα κονδύλια από όσα χρειάζονται. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να φύγουμε από αυτή την αίθουσα έχοντας μια συγκεκριμένη ιδέα για το τι ακριβώς λείπει. Ξέρουμε ότι είναι ανεπαρκής ο προϋπολογισμός και θα ήθελα με πλήρη συνείδηση να πάρω την αποφασή μου. Νομίζω ότι δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας και σε περίοδο κρίσης θα πρέπει να λέμε τι χρειαζόμαστε. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε διάφορες περιπτώσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε επίδειξη φαντασία σε ό,τι αφορά τα μέσα. Σε διεθνές επίπεδο υπάρχει η πρακτική των special drawing rights εάν υπάρχει μια περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα κονδύλια η περίοδο προετοιμασίας του προπολογισμού θα μπορούσε να υπάρχει το αυτοδικαίωμα αυτό για μια συγκεκριμένη χώρα βέλος. Νομίζω ότι με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαμε να ε, καταστήσουμε περισσότερο υπεύθυνε τις χώρες που δέχονται ε, πρόσφυγες. Ύστερα υπάρχει το πρόβλημα της ε, αρμοδιότητας. Για ποιο λόγο υπάρχει πρόβλημα, γιατί είναι ένα θέμα διακυβερνητικό. Υπάρχουν, ε, ε, υπάρχει λίγο διακυβερνητικό και λίγο ομοσπονδιακό. Δηλαδή βαδίζουμε με το κεφάλι στον τοίχο και ο συνάδελφος έχει δικαίωμα που λέει ότι δεν είναι μια κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι η κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν δεν αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Δεν θα μπορούν να δώσουμε ένα πρόσωπο σε αυτή την πολιτική, γιατί δεν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να υπάρξει ένα συντονιστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα πολιτικής ε, προστίγων. Χρειάζεται ένας ηγέτης εσείς κάνετε μια άψογη δουλειά, δεν, ε, πραγματικά δεν θέλω να σας κρίνω για τίποτα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένας γνωστός πολιτικός υπεύθυνος, ο οποίος να έχει κάποια εξουσία, η οποία θα πρέπει να αναδύεται, να, να, πρέπει να προκύψει από το Βριανό συμβούλιο. Διαφορετικά πιστεύω ότι πάμε κατευθείαν για να χτυπήσουμε το κεφάλι μας ε, στον τοίχο. Χρειάζεται λοιπόν ε, κάποια ε, διαφάνεια και ορισμένες προτάσεις σχετικά με το θέμα της διακυβέρνησης. Οι χώρες μέλη δίνουν μια αξιολέπητη εικόνα. Θα μπορούσαμε να καθέσουμε τώρα ερώτημα ποια είσαι Ευρώπη, μας ικανοποιεί αυτή η κατάσταση. Πραγματικά ντρεπόμαστε να βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να γίνουμε συνεργοί σε αυτή την αδυναμία ενώπιον ενός προβλήματος που μας αφορά όλους. Ευχαριστώ πολύ. Δύο διευκρινήσεις θα ήθελα μόνο. Αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει 4 δισεκατομμύρια από την αρχή της ανθρωπιστικής κρίσης και ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν συγκεντρώσει μόνο το 33% των κονδυλίων που χρειάζεται. Οι Ηνωμένε Πολιτείε από την άλλη κάνουν περικοπές. Μπορούμε να μάθουμε τι συμβαίνει ακριβώς εκεί. Πολλά ε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πολλοί πολίτες κιόλα μα ρωτούν γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείες δεν συμμετέχουν στην ε, βοήθεια της ε, κρίσης αυτής. Έπειτα, όπως είπε και η Χέιντι Χάουταλα, το πρόβλημα του να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια. Έχω να πω ότι όταν πήγαμε στην Τουρκία, Είδαμε πάρα πολλούς εκτοπισμένους ανθρώπους και φυσικά μην ξεχνάμε και τους εσωτερικά εκτοπισμένους. Στη Συρία είναι περίπου 6,5 εκατομμύρια πολίτες. Όταν λοιπόν πήγαμε στην Τουρκία ακούσαμε ότι το 83% της ανθρωπιστικής βοήθειας πηγαίνει στην Νότσα, στη Δαμασκό, όμως δεν μπορούν να ε, κάνουν τίποτα μετά από εκεί, δεν μπορούν να βγάλουν κόσμο. Υπάρχουν προβλήματα στα σύνορα, δυσκολία στην μετακίνηση και τα χρήματα για την ανθρωπιστική βοήθεια δεν φτάνουν ε, πέρα από τη Δαμασκό διότι ε, υπάρχουν διάφορα, διάφορα κολλήματα εκεί. Ε, κύριε Βέντα, κάτι θέλετε να πείτε γι' αυτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι περισσότερες παρατηρήσεις και ερωτήσεις ήδη διατυπώθηκαν για τα συστήματα, για την παροχή βοήθειας, για τα θέματα της Ανατολικής Ουκρανίας και των συνόρων προς τη Ρωσία. Υπάρχει πρόβλημα εδώ να φτάνει η ανθρωπιστική βοήθεια επιτόπου και τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν για το πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε, να συνδράμουμε, να συνδράμουμε τα αιτήματα αυτών των ανθρώπων. Αναφέρθηκε πιο πριν η Συρία, η Εμένη, και τα μεταναστευτικά ρεύματα εξ Ανατολής, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά και πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε δράση για την παροχή βοήθειας στην προέλευση ακριβώς, στην απαρχή των ρευμάτων αυτών των προσφύγων προς την Ευρώπη. Μάλιστα λοιπόν, έχετε να απαντήσετε σε πολύ δύσκολα ερωτήματα, αλλά η κύρια ερώτηση είναι αν υπάρχουν αρκετά ευρωπαϊκά κονδύλια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα ερωτήματα αυτά. Πιστεύω ότι όλοι μας συμφωνούμε με την ανάλυση της κατάστασης και ο κύριος Γκερέρο και όσοι πήραν το λόγο κατέστησαν σαφές ότι Κοινοβούλιο και Επιτροπή συμπλέουν. Αν είχα μια μαγική λύση για να υποχρεώσω τις ε, ε, χώρες μπέλη να κάνουν κάτι, να το έκανα. Ε, στα γαλλικά λέμε ότι ακόμα και το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο δεν μπορεί να δώσει τίποτα περισσότερο από όσα έχει. Πώς μπορούμε να υποχρεώσουμε τις χώρες μέλη. Τι να σας πω, ειλικρινά δεν ξέρω. Προσπαθούμε να τις ε, πείσουμε. Ο πρόεδρος Γιούνκερ εδώ και δέκα μέρες ήρθε και σας μίλησε και πραγματικά μίλησε για περισσότερη ευρωπαϊκή ε, αλληλεγγύη Γίνονται διαρκώς προσπάθειες. Ο πρόεδρος Τούσκ συγκάλεσε για αύριο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πέρα από αυτό, τι να πω, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και ζητάμε περισσότερη αλληλεγγύη από όλους συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών. Εμείς σε επίπεδο προϋπολογισμού, γιατί είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα, σε επίπεδο προϋπολογισμού ξέρετε ότι έχουμε περίπου ένα δισεκατομμύριο το χρόνο, αυτό το προϋπολογισμό, τον χρησιμοποιούμε όσο καλύτερα. Γιατί κάθε χρόνο προσπαθούμε να βρούμε επιπλέον κονδύλια και σήμερα και φέτος ζητήσαμε μία περαιτέρω ενίσχυση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Κάποιος ζήτησε να μάθει τι θα πρέπει να γίνει τον προπολογισμό, να τον τετραπλασιάσουμε, να τον πενταπλασιάσουμε. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να βρεθεί μία πολιτική λύση το πρόβλημα. Ε, οι άνθρωποι που εγκαταλείπουν αυτές τις χώρες το κάνουν γιατί πιστεύουν ότι η Ευρώπη είναι Ελντοράντο. Αυτό είναι το θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Αυτός είναι ένας άλλος ε, τομέας ε, που δεν είναι της αρμοδιότητάς μου. Πιστεύω ότι σε επίπεδο ανθρωπιστικής ε, βοήθειας θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά. Η ανθρωπιστική βοήθεια θα, θα πρέπει να α, μας οδηγήσει στην ενίσχυση οργανώσεων. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα στην Ευρώπη, στις χώρες μέλη. Με οι κρίσεις ε, είναι όλο και περισσότερες. Κρίμα που δεν μπορώ να σας δείξω ένα πίνικα για να δείτε το πώς εκθετικά αναπτύσσεται η κρίση. Δεν έχουμε τίποτα στη διάθεσή μας ή αυτά που έχουμε ε, δεν αρκούν. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Η θα ήθελα να επαναλάβω για μία ακόμα φορά αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια πηγαίνει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να συμβάλλουμε στα ταμεία των χωρών μελών ε, για θέματα που είναι αρμοδιότητας δικής τους. Πέρα από αυτό, θα μπορούσε να υπάρξει ε, να γίνει μία προσπάθεια, αλλά βεβαίως αυτό δεν μπορεί να καλύψει τις ευθύνες των κρατών μελών οι οποίες ε, δεν θέλουν να μοιραστούν όλε όλες αυτές ε, τις ε, αρμοδιότητες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο επιτροπής. Τώρα, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και στην παρέμβαση μου δεν μίλησα γι' αυτό, αλλά θέλω να πω δύο λόγια. Δημιουργούμε αυτό που ονομάζουμε closed funds. πιστεύματα για την Συρία Για τη Συρία δόθηκαν 40 ε, εκατομμύρια ευρώ, 3 εκατομμύρια για την Ιταλία, 5 από τη Γερμανία. Έχετε μία ιδέα λοιπόν γιατί μιλάμε. Τα κάνουμε και πάλι μία έκπληση στις χώρες μέλη για να μπορέσουν να συμβάλλουν το ίδιο και για το ε, Σαχέλε προτάθηκε να δημιουργηθεί ένα ταμείο για το ε, Χέλε Περιμένουμε το ταμείο, για το ταμείο αυτό να κάνουν κάτι χώρες μέρη. Το πλεονέκτημα αυτού του καταπιστεύματος είναι ότι επιτρέπει μια, μεγαλύτερη, ε, μια ευρύτερη χρήση των μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υπάρξει ένας μηχανισμός γρήγορης χρηματοδότησης. Αυτό δεν ισχύει με το Ταμείο Βοήθειας στην Ανάπτυξη. Μετά έχουμε τα ταμεία για τη μετανάστευση που είναι διαρθρωτικά ταμεία και που έχουν ένα πιο δύσκολο, πιο δίσκαμπτο σύστημα. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε κάτι και σε αυτό το σημείο. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε και με τους εταίρους μας της Γενικής Διεύθυνσης σε μια προσπάθεια να βρούμε τους μηχανισμούς που θα μας επιτρέψουν να δράσουμε το συντομότερο δυνατό και πιστεύω ότι εκεί η συνεργασία πάει καλά. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία και την Σερβία, για την Σερβία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού υπήρξε μια ενίσχυση 1,8 εκατομμύρια ευρώ για τη Σερβία. Δεν είναι πολύ μεγάλη ενίσχυση, αλλά θελήσαμε να δώσουμε ε, χρήματα σε οργανώσεις όπως το World Food Program της ε, ΜΚΟ για να υπάρξει ε, περίταλψη. Βεβαίως δεν είμαστε εκεί για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Προσπαθούμε να κινηθούμε στα πλαίσια του δυνατού σε ό,τι αφορά την Τουρκία και η Τουρκία είναι μια διαφορετική περίπτωση. Η Τουρκία έχει ένα αρκετά μεγάλο προϋπολογισμό στα πλαίσια τα προ, προενταξιακά. Το θέμα είναι πώς να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά με κονδύλια για την ε, προσχώρηση, με δράσεις ευρύτερης κλίμακας, τον τομέα πούμε της εκπαίδευσης. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσα από αυτό το καταπίστευμα. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι. Από πού προέρχονται τα χρήματα, από το προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το κεφάλαιο 4. Πώς θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να σκεπτούμε στα πλαίσια της αναθεώρησης των ε, οικονομικών προοπτικών. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα για να έχουμε την βεβαιότητα ότι θα μπορούμε να αντιδρούμε περισσότερο έγκαιρα σε ό,τι αφορά τα σημεία, τα θέματα αυτά. Πώς ε, να υποχρεώσουμε την Ελλάδα να θέσει σε εφαρμογή το μηχανισμό. Τι να πω. Θα μιλήσω αύριο με τον διευθυντή μου, θα ήθελα να του υπενθυμίσω ότι υπάρχει ο μηχανισμός, η ενίσχυση που δεν φτάνει στους αποδέκτες και εκεί προσπαθούμε να αναπτύξουμε έναν διάλογο και ο Επίτροπος Αβρομόπουλος με τον Επίτροπο Στυλιανίδη θα πάνε σύντομα στην Τουρκία για να εξετάσουν ορισμένα θέματα μαζί με τις αρχές έτσι ώστε να έχουν τη βεβαιότητα ότι η ενίσχυση θα φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει σε ό,τι αφορά την ενίσχυση προς τη Συρία. Προσπαθούμε να έχουμε την ε, βεβαιότητα ότι η ενίσχυση αυτή θα φτάσει στον προορισμό της Και πάλι προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε και πάρα πολλές δυνατότητες. Σε ό,τι Α, Ουκρανία. Σε ό,τι αφορά την ε, Ουκρανία, Έχουμε ξεκινήσει κάποια συζήτηση και με τη Ρωσία και με τις Ουκρανικές αρχές γιατί μέχρι το μέσο της χρονιάς η δυσκολία πρόσβασης οφείλεται στις αρχές της Ουκρανίας. Τώρα το πρόβλημα έχει ρυθμιστεί προσπαθούμε με τη Μόσχα να διευκρινίσουμε αυτή την κατάσταση και προσπαθούμε να θα ήθελα να στείλω το μήνυμά σας στον κύριο Κρίς Εδώ βεβαίω έχουμε να κάνουμε με θέματα μεταναστευτικά, για τα οποία είναι ένας άλλος επίτροπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αλληλεγγύη σα. Πιστεύω ότι κινούμεθα προς την ίδια κατεύθυνση. Ξέρω ότι και ξέρω ότι πάντοτε μπορώ να υπολογίσω στη βοήθειά σας. Ναι, πιστεύω πως αν αθροίσουμε όλα τα χρήματα που έχουν διαθέσει τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την κρίση στα σύνορά τους, θα συνειδητοποιήσουμε ότι θα ήταν ε, πολύ πιο χρήσιμο να τα διέθεταν για ανθρωπιστική βοήθεια επιτόπου στις περιοχές ε, που υφίστανται κρίσεις. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ και ελπίζω να σας ξαναδούμε όχι σε πλαίσιο κρίσης πάλι. Λοιπόν, συνάδελφοι, η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου και τις 13 Οκτωβρίου. Θα ήθελα μόνο να πω, να σημειώσετε ότι ενδεχομένω να συνεδριάσουμε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Θα είναι μία έκτακτη συνεδρίαση, ειδική συνεδρίαση όπου θα μας κάνει μία παρουσίαση η Φεντερίκα Μογκερίνη και ο Επιτροπος Μίμητσα για τη Συμφωνία του Κοτονού για τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων, τη συμφωνία του Κοτονού. Να σα ενημερώσω λοιπόν από τώρα ότι ενδεχομένω να συνεδριάσουμε τότε. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Θα επανέλθουμε με τους συντονιστέ σε λίγο.